Meine Κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση, συνεχίζεται η ψηφοφορία με την έκθεση Gross για τις εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές. Έχουμε 42 τροπολογίες της Επιτροπής Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δέκτη. Ο κύριος Κάμπελ. Κύριε Πρόεδρε, δεν μου δόθηκε ο λόγος νωρίτερα. Θεωρώ ότι η ελεύθερη κυκλοφορία